Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ πολύ. Συνεδριάζουμε σήμερα για να συζητήσουμε δύο εκθέσεις. Έκθεση πρωτοβουλίας Κατραχάσα και, μια... και ένα σχέδιο νομοθετικής έκθεση στη συνέχεια. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση όσον αφορά τις τροπολογίες και για τις δύο αυτές εκθέσεις. Έχουμε 499 τροπολογίες για την νομοθετική έκθεση FC2 όπου έχουμε 51 τροπολογίες για το σχέδιο έκθεσης και 315, 395 τροπολογίες όσον αφορά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Σας δόθηκαν στις τελευταίες ημέρες διαφορετικές εκδοχές. Θα γίνουν και συνεδριάσεις στο μέλλον των ε, σκιωδών εισηγητών, ήδη την εβδομάδα στο Στρασβούργο και προβλέπεται και μία συνεδρία στο σχεδόν συγητών την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Σας υπενθυμίζω το Συμβούλιο έχει ήδη καταλήξει σε μία τοποθέτηση για το FC2 το Δεκέμβριο του 2016. Καταρχάς όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε παρατηρήσει για την μερίσια διάταξη, αν μπορούμε την εγκρίνουμε ως έχει. Ρομπέρτο, έχεις να κάνεις παρατηρήσεις. Ας δώσουμε τότε το λόγο ευθύ αμέσω στους δύο συνεισηγητές μας. Καταρχάς ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να διευθετήσουμε. Συμφωνείτε να εξετάσουμε τις τροπολογίες και για τις δύο αυτές εκθέσεις από κοινού. Γιατί αν είναι να δούμε ξεχωριστά πρώτα δηλαδή την νομοθετική έκθεση και την έκθεση πρωτοβουλίας, τότε ενδεχομένω να μην καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή μέχρι τις 8. Συμφωνούν λοιπόν οι συνεισηγητές να εξετάσουμε από κοινού τι τροπολογίε και για τις δύο εκθέσει. Συμφωνούμε πολύ ωραία. Ωραία, θα ξεκινήσει πρώτος, ο Ούντο Μπούλμαν, παρακαλώ. Äh, Ευχαριστώ τους ε, συμπροέδρους. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους ε, για το μεγάλο ενδιαφέρον και για τις δύο εκθέσεις. Ε, συγκεκριμένα έχουμε 395 τροπολογίες ε, για την εφαρμοστική έκθεση και 499 για την νομοθετική πρόταση. Αυτό σημαίνει ότι ακριβώς οι συνάδελφοι θέλουν εντατικά να συμμετάσχουν και αυτό είναι καλό. Σήμερα, ο Χωσέ Μανουέλ και εγώ ε, θα ακούσουμε προσεκτικά. Θέλουμε να να δράξουμε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε με τους συναδέλφους, να μάλλον να ακούσουμε τους συναδέλφους, να ακούσουμε τις προτάσεις τους για να μας πούνε συνολικά πώς βλέπουν ε, αυτή την έκθεση για να μπορέσουμε να έχουμε την συνολική μας διατύπωση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες αντιφάσεις σε σχέση με την εφαρμοστική έκθεση η οποία επικεντρώνεται πολύ στις αιτιολογικές σκέψεις. Υπάρχουν πολλές προτάσεις που έγιναν για τη βελτίωση αυτών και έχουμε βρει και κάποιες συμβαστικές τροπολογίες για κάποιες από αυτές που έχουν προταθεί. Είναι μάλιστα σε έγγραφη μορφή και ζητήσαμε μέχρι αύριο στις 2 το μεσημέρι να λάβετε θέση να πείτε τι πιστεύετε για αυτές τις τροπολογίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρως διαφανή και υπεύθυνη διαδικασία με τη δική σας συνεισφορά και την Τετάρτη ε, να συναντηθούν οι σκιώδεις. Για την νομοθετική έκθεση, την έκθεση νομοθετικού περιεχομένου, συνολικά υπάρχουν κάποια βασικά σημεία στα οποία θα επικεντρωθεί η, συζήτηση. Να τα αναφέρω γιατί θεωρώ ότι πρέπει ε, να κάνουμε πολύ καλή συζήτηση μεταξύ μας για αυτό το θέμα. Χρειάζεται ένα θέμα είναι οπωσδήποτε το θέμα του earmarking και οι δύο συνεισηγητές ε, πρότειναν να πάμε πέρα από την πρόταση της Κομισιόν και συνολικά ε, στα ε, πεδία εφαρμογής του FC2 να έχουμε ως κριτήριο τους στόχους ε, αηφορίας και βιωσιμότητας των Ηνωμένων Εθνών. Ουσιαστικά αυτό εν μέρη μπορεί να γίνει αποδεκτό, από την άλλη στην ουσία δείχνει και στους συναδέλφους Ποια είναι η αρχική πρόταση της Κομισιόν, το 14% COP21. Είναι οι στόχοι που θέλουν, θέλουμε να ενταχθούν. Υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο, η προσθετικότητα, η έννοια και η εκτέλεση της προσθετικότητας. Εδώ πρέπει το κόπορτ να είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο και υπάρχουν διάφορες απόψεις που έχουν ε, να κάνουν με τον ορισμό του Special Operations. Πώς ε, ε, δηλαδή το θεωρούμε από την πλευρά των ευρωπαϊκών επενδύσεων. Πρέπει να το συζητήσουμε για τη διακυβέρνηση, governance, αυτό είναι το τρίτο μου σημείο. Υπάρχουν και εκεί προτάσεις από τους συνεισηγητές να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία πιο στοχοθετημένη, να υπάρχει μια σωστή παρακολούθηση από το Κοινοβούλιο και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε πώς θα το επιτύχουμε. Επίσης, βλέπω ότι η διαφοροποίηση προς ε, τομεακές και γεωγραφικές συνιστώσεις είναι πολύ σημαντική. Αναφέρεται σε όλες τις ε, ε, τροπολογίες και τις απαιτήσεις των συναδέλφων. Αυτό που λέει κύριος ο Χωσέ Μανουέλ, αυτό το θέμα που μόλις σας είπα, είναι αυτά, αυτά τα θέματα που έθιξε έχουν να κάνουν με τη δική μου δουλειά σα, που σας παρουσίασα. Ωραία. Οπότε γίνεται και έτσι η μετάβαση στον Χωσέ Μανουέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφερόμαστε, όπως είπατε και εσείς, στις δύο εκθέσεις, στην πρόταση κανονισμού, καθώς επίσης και στην πρόταση για την εφαρμογή του ΕΦΣΥ. Θα πρέπει οι δύο αυτές εκθέσεις να συνδυαστούν, να κινηθούν παράλληλα, γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε τελικά να δικαιολογήσουμε και την παράταση της διάρκειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Ευχαριστήσω καταρχάς τους και οδησηγητές για τις τροπολογίες τις οποίες κατέθεσαν και να ευχαριστήσω προφανώς και τον συνάδελφο Μπούλμαν για την εργασία που κάναμε από κοινού προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων που θα λειτουργεί πραγματικά υπέρ της κοινωνικής, εδαφικής συνοχής και οικονομικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει το Ταμείο αυτό να μπορεί να επωφελεί όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπαμε ότι δεν πρέπει εδώ πέρα να θεσπίσουμε ποσοστώσεις αυτό είναι σαφές. Θα πρέπει να προωθήσουμε σαφώς την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει όλα να γίνουν μόνο στο σκέλος της ζήτησης. Αυτές οι ευρωπαϊκές πλατφόρμες επενδυτικές αλλά και ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών δεν αξιοποιούνται πλήρως από τα κράτη-μέλη. Οι συμβουλές όμως που δίδονται από τον κόμβο αυτό είναι δωρεάν και είναι πάρα πολύ σημαντικές, κρίσιμες, καθοριστικές θα έλεγα συμβουλές αυτές, προκειμένου να ολοποιηθούν επενδυτικά προγράμματα ποιότητας, προκειμένου να υποβληθούν τα προγράμματα αυτά και προκειμένου να μπορούν να λειτουργούν ομαλά οι επενδυτικές πλατφόρμες. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να έχουμε διεθνικά, διασυνοριακά ή διαφορετικά τομεακά προγράμματα και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να έχουμε πλατφόρμες οι οποίες θα προωθήσουν και προγράμματα, έργα μικρότερους και, μικρότερης κλίμακας, μικρότερου μεγέθους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το ταμείο αυτό να είναι ανοιχτό προς όλες τις επενδυτικές προτάσεις, ακόμα και στις πιο μικρές, και το ταμείο αυτό θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ε, τοπική πραγματικότητα που ισχύει για κάθε σχέδιο το οποίο έχει υποβληθεί. Και να ληφθεί υπόψη επίσης και το ζήτημα της προστατικότητας. Να γνωρίζουμε δηλαδή ποιες επιπτώσεις, εποφελής ή μη, μπορεί να έχει υλοποίηση ενός σχεδίου. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι το ΕΦΣΙ δεν είναι αρκετά προβεβλημένο. Το σκέλος του ΕΦΣΙ που έχει να κάνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι όντως πάρα πολύ ε, σημαντικό και γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία. 400.000 περίπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατάφεραν να αποφεληθούν από το ΕΦΣΥ. Έχουμε και την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Υποστηρίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πολύ συχνά δεν γνωρίζουν όμως ότι μιλάμε για ένα πραγματικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να προωθήσουμε και να προβάλλουμε περισσότερο το ΕΦΣΥ. Όσον αφορά την διακυβέρνηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή να διέπεται από απόλυτη διαφάνεια. Όταν μιλάμε λοιπόν για διακυβέρνηση, ουσιαστικά αυτό που εννοούμε είναι ότι οι αποφάσει που λαμβάνονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη, από του παρεμβαίνοντε, σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να δικαιολογούνται απόλυτα και πλήρω. Πόσο μάλλον που μιλάμε αυτή τη στιγμή για πολύ ευαίσθητε πληροφορίε. Η γεωγραφική διαφορετικότητα και αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη Κάθε φορά που αναφερόμαστε στον ε, συγκεντρωτικό αυτό χαρακτήρα που θα πρέπει να έχει το πρόγραμμα αυτό και όταν αναφερόμαστε στο ότι θα πρέπει να προωθεί το πρόγραμμα συνοχής. Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και στην, ε, στα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα ταμεία αυτά δεν αντικαθιστούν το ένα το άλλο. Μπορεί όμω να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, μπορεί να λειτουργήσουν συνδυαστικά. Επίση, είναι πολύ σημαντικό οι υποχρεώσει που έχουν ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δεσμεύσει όσον αφορά τι κλιματικέ αλλαγέ, θα πρέπει και αυτέ να ενσωματωθούν στη στρατηγική του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα αναφερόμαστε σε μία οριζόντια δέσμευση που επηρεάζει όλα τα επενδυτικά προγράμματα. Στο μέτρο λοιπόν του δυνατού θα πρέπει η κλιματική αυτή διάσταση να είναι παρούσα σε όλα τα προγράμματα, σε όλα τα έργα τα οποία υποβάλλονται για έγκριση. Έπειτα, πέρα από την κλιματική διάσταση έχουμε και την κοινωνική διάσταση. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ένα 4 μόνο της 100, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση των υποδομών, έχουμε, έχουμε λάβει υπόψη την κοινωνική διάσταση ενδεχομένως το ποσοστό αυτό να πρέπει να αυξηθεί. Επίσης, έχουμε σημαντικές επενδύσεις στον κοινωνικό τομέα, οι οποίες θα πρέπει να αυξηθούν καθότι είναι καθοριστική σημασία για την Ευρώπη. Όταν μιλάμε και οικονομική, εδαφική, κοινωνική συνοχή, προφανώς αυτός είναι ένας ευκταίος στόχος, ο οποίος θα πρέπει να χαρακτηρίζει όλες τις πτυχές του Ταμείου αυτού. Το Ταμείο αυτό έχει ήδη οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Είναι επίσης ένα ταμείο το οποίο έχει υποστηρίξει τις επιχειρήσεις, όπως σας το είπα, και είχε και θετικές επιπτώσεις όσον αφορά τον ίδιο τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφίσταται παρόλα αυτά όμως ένα χάσμα επενδύσεων Συντοποιούμε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν αποτελεί πανάκια. Εξακολουθούν και υφίστανται εμπόδια στι επενδύσει. Θα πρέπει εμεί να καταρρύψουμε τα εμπόδια αυτά, προκειμένου οι επενδύσει να μπορούν να λαμβάνουν χώρα ομαλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το καθήκον μα. Ευχαριστούμε πολύ. Α δώσουμε τώρα το λόγο στου σκιώδει εισηγητέ. Σα παρακαλώ πολύ, μην μιλήσετε πάνω από δύο λεπτά. Το λόγο λοιπόν έχει ο κύριο Κάρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω από την έκθεση ίδια πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι είναι ισορροπημένε οι συμβαστικέ προτάσεις. Νομίζω καλύπτουν τις διάφορες ομάδες. Δύο πράγματα θα ήθελα να αναφέρω ακόμα. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα κριτήρια των έργων δεν επιτρέπεται να χαλαρώσουν ούτε στο θέμα του στόχου των επενδύσεων των 350 ε, 450 εκατομμύρια, ούτε για το θέμα της ε, διαφοροποίησης για να κλείσουμε διάφορες ε, τρύπες και κενά στην Ευρώπη. Γιατί χρειαζόμαστε ισχυρά διαρθρωτικά μέτρα. Στο θέμα της νομοθεσίας, στο νομοθετικό τμήμα, Κάποιες ε, τροπολογίες της ομάδας μου υπενθυμίζουν ότι κάποιες ε, θέσεις χρηματοδότησης δεν ενδείκνυνται για όλα τα έργα και ταυτόχρονα βεβαίως οι διατάξεις της εγγύησης ε, του Ταμείου δεν επιτρέπεται να δημιουργούν στρεβλώσεις της αγοράς. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται συζήτηση για τον, για τον ορισμό των διασυνοριακών έργων με τρίτες χώρες, το άρθρο 8. Η Επιτροπή μέχρι τώρα τους ή άλλως δεν έχει υποβάλει τέτοια έργα, κάτι το οποίο βεβαίως δεν είναι προς το συμφέρον μας ως ε, νομοθέτες. Θέλουμε λοιπόν περισσότερη διαφάνεια. Και Βεβαίω θέλουμε περισσότερες αποστολές για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Συμβουλών ε, Επενδυτών. Και βεβαίως να υπάρξει μια γεωγραφική ισορροπία και να ενισχύσουμε συνοριακά τις ε, πλατφόρμες. Θα ήθελα λοιπόν ε, να πω πως υπάρχουν ακόμα τα 7 αυτά σημεία τα οποία λείπουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έντερ Γκάρδια Σάμπαλ. Δεν τον βλέπω. Και ποιος θα μιλήσει. Θα δώσω τον λόγο στον Σάντερ Λούνες, δεν είναι εδώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκπροσωπήσω το ΙΣΙΑΡ και ιδιαίτερα τον συνάδελφο Λούνς, ο οποίος δυστυχώς κολλείεται. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν, αλλά να αναφερθώ σε κάποια σημεία κριτικής ε, που βλέπουμε ως ECR στην παράταση του FC ως FC2. Θεωρώ ότι συμφωνούμε. Το FC ε, δεν είναι πανάκια. Δεν μπορούμε να γυρνάμε από εδώ και από εκεί και να θεωρούμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα λύσει όλα τα οικονομικά προβλήματα της Ένωσης. Για εμάς αποφασιστικό λοιπόν είναι το ερώτημα γιατί μιλάμε τώρα ήδη για το FC2 όταν δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί το πρώτο FC. Ειδικά δεδομένου του ότι στο FC2 δεν φαίνεται να λειτουργεί όπως ε, το θέλαμε. Παρά το όσα λένε μερικοί συνάδελφοι, αποδείξεις δεν υπάρχουν. Και δεν ε, είναι δυνατόν βεβαίως ε, να έχουμε ένα ανταγωνισμό με υφιστάμενα προγράμματα. Θα υπάρξουν λοιπόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού γιατί οποιοδήποτε συμμετέχει στο ΕΦΣΥ θα είναι σε καλύτερη θέση από κάποιον ο οποίος δεν συμμετέχει. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα λοιπόν λέμε εμείς ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να αποφασίσουμε για ένα δεύτερο στρατηγικό ταμείο επενδύσεων. Και αν μιλήσουμε επί της αρχής πρέπει να διασφαλίσουμε να υπάρχει προσθετικότητα, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και την γεωγραφική πτυχή, γιατί υπάρχουν οπωσδήποτε διαφορές στο πού θα με το ΕΦΣΥ. Και εδώ πέρα υπάρχουν παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι δεν είναι επιτυχημένο. Όταν παραδείγματο χάρη είναι στην Γερμανία, ε, χρηματοδοτούνται δημόσια έργα στα οποία ενώ, με συγχωρείτε, το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να δανείζεται με αρνητικά επιτόκια. Ε, δεν χρειάζεται το ΕΦΣΙ λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο Ραμόν Τρεμόσα Μπαλσέτς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε δύο λεπτά βλέπω ότι υπάρχουν εδώ πέρα εκατοντάδες τροπολογίες και πολλές από αυτές αφορούν το τι είναι ένα επιπρόσθετο έργο και τι έργα πρέπει να χρηματοδοτεί το ΕΦΣΙ και τι όχι. Αυτό είναι καλό σημάδι νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε για τους τελικούς ε, χρήστες που έχουν δεσμευτεί ε, εξ ονόματος του ΕΦΣΙ. Νομίζω είναι καλή αυτή η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Επίσης ε, βλέπουμε ότι υπάρχει συγκέντρωση έργων στις ίδιες περιφέρειες για λόγους πολιτικούς και όχι οικονομικούς. Ο τρόπος για να λυθεί αυτό είναι να έχουμε μια καλύτερη σχέση μεταξύ του ΕΦΣΙ και των τοπικών επενδυτικών τραπεζών, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται καλύτερα η χρηματοδότηση. Και τέλος, πρέπει να υπενθυμίζουμε στους ευθύους μας ότι το ΕΦΣΙ πρέπει να χρησιμοποιείται για να ε, έχει κάποια προσθεμένη αξία. Όχι τα ίδια και τα ίδια. Δεν έχουμε και κάποια μανία με, για τη γεωγραφική κατανομή. Δεν είναι ταμείο συνοχής. Πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην αποτελεσματικότητα και την προσθέμενη αξία και να δούμε ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για να τα επιτύχουμε αυτά. Γιατί υπάρχουν και άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια για να επιτύχουμε τη γεωγραφική ισορροπία. Τέλο, για τη δική μου την περιφέρεια. Λοιπόν, ε, θα πρέπει να προσέξουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην ε, τελικά βρεθεί πίσω από τις αποφάσεις κάποιων ε, κυβερνήσεων που θα αποφασίζουν με άλλα κριτήρια. Τα κριτήρια δηλαδή που θα αποφασίσουμε εδώ να μην τα αλλάξουν στις πρωτεύουσες για να κάνουν τα ίδια και τα ίδια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Νίλς Τόρβαλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν Υπάρχουν κάποιες γερμανικές λέξεις που χρησιμοποιούνται και στα αγγλικά. Ε, χερκακία ας πούμε. Αλλά βεβαίως ε, και η λέξη τσουγκσβάγκ. Δηλαδή ότι υπάρχει μια πίεση να προχωρήσουμε. Εδώ είναι χρονική πίεση, το βλέπετε ότι κινούμαστε σε ένα πολύ γενικό επίπεδο και δεν ε, μπαίνουμε στις συμβαστικές προτάσεις. Λοιπόν, κάποιες παρατηρήσεις. Η προσθετικότητα συζητήθηκε πολλές φορές και νομίζω ότι χρειάζεται κάποια διευκρίνηση. Η διαφάνεια επίσης από την αρχή. Και νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια από την Τράπεζα Επενδύσεων. Αλλά πρέπει να πω τώρα ότι δεν μου αρέσει να μπαίνουμε σε τόσο ε, μεγάλες, σε τόσο μικρές με συγχωρείτε, λεπτομέρειες της ε, διαχείρισης ως κοινοβουλίου. αν και αντιλαμβάνομαι ότι χρειαζόμαστε κάποιες διευκρινήσεις για το πώς λειτουργεί το ΔΣ. Γιατί αν λειτουργεί με στόχο το ΠΑΤ που λέμε στο ΣΚΑΚΙ, την ισοπαλία, δεν είναι και ιδανικό. Λοιπόν, Έχουμε και αυτόν τον ε, κόμβο των συμβουλευτικών των επενδυτών, συζητάμε και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι ενδιαφέρουσες και ειδικά όταν συνδυάζονται με τους στόχους για το κλίμα και την τεχνολογία. Πρέπει αυτά να τα συνδυάσουμε. Αν δεν τα συνδυάσουμε, τότε τα πράγματα δεν λειτουργούν. Λοιπόν, τέλειος χρόνος. Με ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ. Εφόσον δεν είναι εδώ ο Φάμπιο Ντεμάση, ο κύριος Βιαγκάσκη. Ευχαριστώ. Υπάρχουν ε, κάποιες πολλές αλλαγές σε αυτή την αρχική κανονισμό, συγκεκριμένα η κατάργηση του άρθρου που υποχρεώνει σε μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ε, του σχεδίου ε, προκειμένου να υπάρξει παράταση. Καταργείται λοιπόν αυτό το άρθρο, άρα θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν τα δεδομένα τα οποία θα μας επέτρεπε να αξιολογήσουμε την ανάγκη, ε, το λόγο που θα υφίστατο για να παρατείνουμε αυτό το σχέδιο. Τα μακροοικονομικά, οι μακροοικονομικές επιπτώσεις σε επίπεδο επενδύσεων δεν αλλάζουν. Επίσης η θεματική και η γεωγραφική συγκέντρωση, η προσθετικότητα είναι θέματα που μας προκαλούν αμφιβολίες. Μιλάω για παράδειγμα για αυτό που συμβαίνει στην Πορτογαλία. Πόσο ξέρω δεν υπάρχουν πραγματικές επενδύσεις. Ε, υπάρχει μόνο ένα έργο που δόθηκε στο Δημαρχείο της Λισαβόνας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, με περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Και, συγγνώμη, 50 ε, εκατομμύρια ευρώ. Αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε αυτό το σχέδιο Juncker για να κάνουμε επενδύσεις στο Δημαρχείο της Λισαβόνας. Μια τέτοια κριτική ας πούμε υφίσταται. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να ζητούμε να υπάρχει πραγματικά ένα δημόσιο σχέδιο επενδύσεων, ένα ε, σχέδιο το οποίο θα προσανατολίζει, θα διοχετεύει τις ε, ιδιωτικές επενδύσεις, θα χρησιμοποιεί τις δυνατότητες ε, των ιδιωτικών επενδύσεων για να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις και όχι στρεβλώσεις. Αυτό που είναι σημαντικό λοιπόν είναι να έχουμε επενδύσει σε ε, υποδομή που θα έχουν τραβήξει ιδιωτικές επενδύσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τους δύο συνεισηγητές. Έχουμε αρχίσει να σχολιάζουμε τις πολλές αυτές τροπολογίες που έχουμε και για τις δύο εκθέσεις και απευθύνομαι στην κυρία Ρουμπιάλ. Θέλετε να πάρετε τώρα το λόγο ή αφού μιλήσουν πρώτα οι υπόλοιποι ομιλητέ. Θα μιλήσετε τώρα. Σας ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε που έφτασα έτσι με καθυστέρηση. Έφτασα λίγο αργότερα από ό,τι προβλεπόταν. Ωστόσο, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και στους δύο εισηγητές και είχα μάλιστα τη δυνατότητα να συνεργαστώ και με τους δύο και για τις δύο εκθέσεις. Τους εύχομαι λοιπόν Καλή επιτυχία με τις 500 τόσες τροπολογίες, Πρόεδρος. Πολύ σωστά τις μετρήσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μυριάντα δεν είναι εδώ πέρα και ούτε την αντικαθιστεί κάποιος. Μπας Εκούτ. Ούτε και αυτός είναι εδώ. Τζόρντι Σόλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι δικές μας τροπολογίες εστιάζονται στα προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει κατά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων στην πρώτη του εκδοχή και οι τροπολογίες μας λοιπόν αυτές ευθυγραμμίζονται και με άλλες κριτικές αξιολογήσεις που έχουν γίνει για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και συγκεκριμένα μετά όσα λέγει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού συνεδρίου, καθώς και αυτό που λένε οι εκθέσεις διαφόρων εξωτερικών ελεγκτών. Θεωρούμε ότι υπάρχουν τρία, τρεις τύποι προβλημάτων. Πρώτον, επίπτωση και διαφάνεια. Θεωρούμε ότι υπάρχουν ελάχιστε αποδείξει αυτή τη στιγμή ότι οι επενδύσεις αυτές είχαν όντως θετικό αντίκτυπο στο κενό παραγωγής και στην έλλειψη θέσεων απασχόλησης. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες ώστε να αποτιμήσουμε πραγματικά τον αντίκτυπο των επενδύσεων αυτών στους τομείς αυτούς και προκειμένου να μπορούμε να κάνουμε κι εμείς πιο ενδελεχή έλεγχο, εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή και το ευρύτερο κοινό. Προτείνουμε ως προς αυτό λοιπόν τις τροπολογίες μας περισσότερο, περισσότερες στι στις εκθέσει. εκθέσεις και μόνο ότι είμαστε υπέρ της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημοσιεύεται ο πίνακας αποτελεσμάτων για τις επενδύσεις αυτές, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνεται αυτό όχι μόνο για τα προγράμματα τα οποία εγκρίνονται, αλλά και τα προγράμματα τα οποία απορρίπτονται. Δεύτερο πρόβλημα, targeting η στόχευση των προγραμμάτων αυτών. Έχουμε επενδύσει πάρα πολύ τελικά στις ε, υποδομές και όχι τόσο πολύ σε μελλοντικές επενδύσεις που θα έπρεπε να γίνουν στα βιώσιμα καύσιμα, για παράδειγμα, ή στις νέες πράσινες μορφές τεχνολογίας. Και νομίζω ότι οι επενδύσεις αυτές πραγματικά δεν έχουν βοηθήσει να καλυφθεί το το επίπεδο φτώχεια το οποίο παρατηρείται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι οι επενδύσει αυτέ θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με, τις στρατηγικές, με του στρατηγικού πολιτικού στόχου Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα 50% των επενδύσεων θα πρέπει να δίνονται σε έργα τα οποία δεν έχουν απλώ μία μα σαφή διάσταση η οποία μπορεί να συνδέεται και με το COP21 αλλά συγκεκριμένα προγράμματα, συγκεκριμένα έργα τα οποία να στοχεύουν στη συμφωνία COP21 και ένα 20% των επενδύσεων αυτών θα πρέπει να βοηθά την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Και τρίτη κατηγορία προβλημάτων, αδυναμιών, το είπαν εκεί οι προαλήσαντες, το ζήτημα της προσθετικότητας. Για μας το σημαντικότερο τμήμα του υφιστάμενου ορισμού για την προσθετικότητα είναι ότι οτιδήποτε δεν μπορεί να γίνει με τα μέσα τα οποία προβλέπονται στο ΕΦΣΥ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε την ευκταία αυτή προσθετικότητα. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε εδώ πέρα την συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία θα πρέπει να συμβάλλει κατά τέτοιο τρόπο στο στην κοινωτική χρηματοδότηση προκειμένου να καταφέρουμε να χρηματοδοτούμε με την συνέργεια Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ΕΦΣΗ συγκεκριμένες ε, πράξεις οι οποίες θα πρέπει να έχουν στρατηγικό χαρακτήρα. Σε αυτό ακριβώς στοχεύει και η δική μας τροπολογία. Τα χρηματοδοτούμε δηλαδή ε, προγράμματα τα οποία θα συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε. Ο Μάρκο Βάλι δεν είναι εδώ είναι και αυτός και ο και για την ΕΚΟΝ και για την Μπάτζα, για το ΕΝΕΦ, Μπάρμπαρα Κάπελ, και αυτή απουσιάζει. Μάρκο ούτε και αυτός είναι εδώ. Πληρώσαμε κατά αυτόν τον τρόπο με τους σκιώδεις συγητές και δίνω την προεδρία στον Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη. Thank Ευχαριστώ. Δεν έχουμε πάρει ακριβώς το αίτημα. αλλά μπορώ να πω ότι μπορούμε να δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν για κάποια σχόλια, κάποια συνεισφορά από την πλευρά της. Κύριος Ρανζέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει μεγάλη σύμπτωση απόψεων μεταξύ της Επιτροπής και των περισσότερων ομιλητών σήμερα. Θέλουμε περισσότερη προσθετικότητα, θέλουμε περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη γεωγραφική ισορροπία. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που θα ήθελα να τονίσω ως προβληματικά εκ μέρους της Επιτροπής. Το πρώτο σχετίζεται με την τιμολόγηση. Προτείνεται στο σχέδιο της έκθεσης ε, το Διευθυντικό Συμβούλιο να έχει την αρμοδιότητα για την ε, τιμολόγηση των πράξεων έψη. Αυτό θα δημιουργήσει νομικό ζήτημα διότι το πρωτόκολλο ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Επενδύσεων που είναι και στη συνθήκη ως ε, προσάρτημα λέει ότι ο διευθυντής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι αυτός που θα θέλει να το, πρέπει να το κάνει αυτό. Επίσης, Τώρα για την ευρωπαϊκή εγγύηση, αν μειώσουμε τις εγγύησεις αυξάνεται το κέρδος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αυτό δεν είναι ο στόχος μας. Δεύτερον, ε, χρηματοδότηση. Όπως γνωρίζετε η Επιτροπή έχει προτείνει να ληφθούν 1,1 δις από το ε, μέσο σαφάς που έχει κανιβαλιστεί από το ΕΦΣΥ. Το Κοινοβούλιο έχει προτείνει το 1,6 δις να μπει στο Connecting Europe Facility, αντί για ένα. Και για τα περιθώρια, από την πλευρά της Κομισιόν έχουμε δυσκολία να αποδεικτούμε βασική αύξηση του περιθωρίου τώρα που έχουμε πιέσει λόγω του Brexit. Είναι δύσκολο να τα συμβιβάσουμε αυτά. Τρίτο σημείο που θέλω να αναφέρω φαίνεται ότι ε, προσπαθούμε να υπάρχει συστηματικό απορτινέσεων προς τον επενδυτή. Είναι λίγο τεχνικό το θέμα, ζητώ συγγνώμη. Είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι το subordination, δηλαδή τα δάνεια ε, μειωμένης εξασφάλισης, είναι πολύ σημαντικό σημείο ε, της ανάληψης κινδύνου, αλλά δεν πρέπει να έχουμε μονίμα αυτό το θέμα. Ε, το να υπάρχει υψηλή εξασφάλιση σε ένα επικίνδυνο project ίσως ε, θα είναι, θα είναι λιγότερο ε, το ρίσκο όταν είσαι ας πούμε μικρότερος εταίρος ε, σε ένα αυτοκινητόδρομο. Πρέπει να έχουμε μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση, να λαμβάνουμε υπόψη μας όλα τα στοιχεία του κινδύνου όπου και να προέρχονται. Τώρα για το COP21. Όπως είπαν κάποιοι ομιλητές από τους Πρασίνους, έχουμε δώσει μεγάλη σημασία. Θέλουμε το COP21 και το σχέδιο επενδύσεων να αλληλοσυμπληρώνονται και να αλληλοενισχύονται. Υπάρχει αυτός ο στόχος του 14% που είναι πολύ φιλόδοξος. Έχουμε πάρει μόνο τα κομμάτια των project που συνεισφέρουν και όχι ολόκληρα τα project υπόψη μας. Επίσης μας ανηχεί λίγο η ιδέα αντικατάστασης με γενική αναφορά στην στόχους της ε, βιώσιμης ανάπτυξης γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν μπορεί να συνεισφέρει σε αυτούς τους στόχους. Βασικά λοιπόν δεν είναι δεσμευτικός αυτός ο στόχος ενώ για το COP21 είναι δεσμευτικός ο στόχος. Τελευταίο σημείο που ήθελα να θέσω αναφέρεται στο σχέδιο έκθεσης. Μιλάμε για την άμεση πρόσβαση των Εθνικών Αναπτυξιακών Τραπεζών στις εγγύησεις, ε, τουλάχιστον στο FC1, η Κομισιόν πριν από ένα χρόνο ανησυχούσε για να είμαστε ειλικρινεί. Θεωρήσαμε ότι αυτή η πρόσβαση θα είναι δύσκολη και δεν υπήρχε και αρκετή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των Εθνικών Αναπτυξιακών Τραπεζών. Σήμερα έχουμε πάνω από 100 project που βασίζονται σε αυτή τη συνεργασία. Στην πράξη λοιπόν αυτό λειτουργεί. Το να ανοίξει αυτή η πρόσβαση στην ουσία δημιουργεί μια σειρά ζητημάτων. Για παράδειγμα, ποιο θα κάνει τη δέουσα επιμέλεια, ποιος ε, θα κάνει τον πίνακα αποτελεσμάτων. Αλλά το πιο σημαντικό είναι δύο μεγάλα ζητήματα που προκύπτουν. Πρώτον, θα ε, επιδεινωθεί η γεωγραφική ισορροπία γιατί δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε. Αν ανοίξουμε πρόσβαση στις Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες, ξέρουμε πολύ καλά ποιες είναι αυτές οι τράπεζες που θα είναι σε καλύτερη θέση να έχουν project. Η SCDC στην Ιταλία, η Κεσδεντεπό στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ισπανία δεν θα είναι οι μικρές, θα είναι οι μεγάλες. Όλη η πίεση λοιπόν που ασκούμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να βελτιώσει τη γεωγραφική ισορροπία θα ε, τεθεί σε κίνδυνο αν ανοίξουμε αυτή την πρόσφαση Και μετά υπάρχει και ένα θολό τοπίο σε επίπεδο λογοδοσίας. Αυτό θα ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο. Για την ΕΤΕΠ μιλάτε στον κύριο Μόιρ στον κύριο Σέρτερελ, να μπορούν να έρθουν αυτοί και να σας πούν τι κάνουν αλλά για το Cash και το ε, ε, ECTP και το KFW ποιος θα έρθει στο Κοινοβούλιο. Για ευρωπαϊκά project είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα πλαίσιο λογοδοσίας σωστό. Αυτό το, το, τώρα που θα πω δεν είναι πρόβλημα, είναι ένα θετικό στοιχείο για το μέλλον. Πολλοί μίλησαν για τη σημασία των κοινωνικών επενδύσεων συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο για να ενισχύσουμε αυτές τις επενδύσεις. Θέλουμε να αυξηθεί σημαντικά η κοινωνική ένταξη και εμπλοκή. Πάνω από το διπλάσιο θα είναι η συμμετοχή χάρη στο ΕΦΣΥ και θα έχουμε και ένα νέο μέσο που θα δώσει πάνω από 3 δις ευρώ επενδύσεων σε μικροδάνεια, μικροεπιχειρήσεις μικροχρηματοδότηση που θα επιφέρει την κοινωνική ένταξη προς όφελος των πολιτών. Έτσι λοιπόν συμφωνούμε με το Κοινοβούλιο ότι οι κοινωνικές επενδύσεις πρέπει να αποτελούν βασική προτεραιότητα. Σταματά εδώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την Επιτροπή και το Διευθυντικό Συμβούλιο. Γιατί και αυτό εκπροσωπείται από όσο ξέρω. Βράτω με τις ευκαιρίες να κάνω κι εγώ ένα σύντομο σχόλιο, δεδομένου ότι υπάρχει χρόνος, για το θέμα της τιμολόγησης. Η δική μου εντύπωση είναι ότι αυτό το κριτήριο του σεβασμού της νομικής ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που από νομική άποψη είναι πολύ σημαντικό αν ακολουθηθεί αυστηρά, θα βρούμε ήδη στοιχεία στον υφιστάμενο κανονισμό, όπου είμαστε κάπως οριακά. Γιατί μιλάμε για ένα πολύ ιδιαίτερο, διαφορετικό οικοδόμημα. Στον κανονισμό ορίζονται υποχρεώσεις σχετικά με το τι ακριβώς αποτελά, αποτελεί νομικά μια απόφαση της ΕΤΕΠ και κάποιους διορισμούς, ας πούμε, που γίνονται. Όλα αυτά τα επιχειρήματα για την ανεξαρτησία της ΕΤΕΠ, κατά τη γνώμη μου, δεν ταιριάζουν πολύ με το τι είναι αυτό το οικοδόμημα στην πράξη. Είναι κάτι βρυδικό. Το βασικό λοιπόν επιχείρημα κατά της τιμολόγησης είναι αυτό το νομικό επιχείρημα γιατί θεωρώ ότι δεν είναι η βάση του πολύ Θεωρώ λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να βρούμε ίσως μια λύση η οποία δεν θα είναι πάντοτε τόσο συμβατή με, την, το καταστατικό της ΕΤΕΠΑ. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να βρούμε μια τέτοια λύση, αλλά Βασίζομαι στην νομική υπηρεσία της Επιτροπής μας ε, ε, ότι θα μας βοηθήσει να πετύχουμε το στόχο που έχει ορίσει ο νομοθέτης για αυτό το σχέδιο. Αυτό είναι το βασικό μου σχόλιο. Σας ευχαριστώ για όλα όσα είπατε. Και τώρα έχουμε την Περβάνς Μπερές στον κατάλογο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αφού ακούσαμε τους εκπροσώπους ε, των δύο αυτών ε, επιτροπών, είναι σημαντικό να μπορούμε να σημειώσουμε πρώτον. Ευχαριστήσω και τους δύο συνεισηγητές. Αποτελεί το κείμενό τους, τα κείμενά τους, πολύ καλή βάση για τη μελλοντική εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να επιμείνω σε τρία σημεία. Πρώτον, Μέσω της παρέμβασής μου αυτής, καταρχάς θα ήθελα προφανώς να υποστηρίξω τις τροπολογίες που έχω καταθέσει. Πρώτον, λοιπόν, όταν είχαμε την έκθεση αξιολόγησης μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι ε, υφίστανται ακόμα κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά την μακροοικονομική επίπτωση που θα έχει η πρώτη εκδοχή του ΕΦΣΥ. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια του ΕΦΣΥ 2 να έχουμε μία γενικότερη στρατηγική ανάκαμψη των επενδύσεων η οποία θα έχει ένα πιο μακροοικονομικό χαρακτήρα. Δεύτερον, το ζήτημα των κοινωνικών επενδύσεων. Άκουσα αυτά του είπε ο Μπέζα ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμφωνώ μαζί του. Ωστόσο, πέρα από τα επιχειρήματα αυτά, ακριβώς με τον τρόπο που ανησυχούμε για να δούμε αν θα καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτοκινητοδρόμους ή όχι, νομίζω θα ήταν χρήσιμο να στείλουμε και ένα παράλληλο μήνυμα, λέγοντας δηλαδή προς τα έξω ότι θα ήταν πολύ καλό να χρηματοδοτήσουμε υποδομές στον κοινωνικό τομέα, δηλαδή νοσοκομεία και σχολεία. Γιατί όλοι μας λένε ότι οι τρεις τομείς οι οποίοι χρηματοδοτούνται πολύ καλά αυτή τη στιγμή και εύκολα από το ΕΦΣΥ είναι ουσιαστικά η ενέργεια, οι μεταφορές και ο ψηφιακός τομέας. Αλλά δεν βλέπουμε να χρηματοδοτούνται πάρα πολλά έργα τα οποία έχουν να κάνουν με σχολεία και με νοσοκομεία. Και τρίτον, το ανέφερε αυτό και ο πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι συνεισηγητές, και συμφωνώ εδώ πέρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαι και πιο φιλόδοξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σαφώ είναι πάρα πολύ θετικό να καλύπτουμε τα πάντα και να καλύπτουμε επίση και του στόχου των μένων εθνών και του στόχου τη COP21. Πολύ καλό όλα αυτά αλλά νομίζω ότι θα είναι καλό να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι. Ακριβώ όπω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ορισμένοι εξημών τουλάχιστον, θελήσαμε να προωθήσουμε το FC1, έτσι και τώρα όταν βλέπουμε πώ έχει κατάσταση στην πραγματικότητα, νομίζω ότι ο στόχο του 50% Α δούμε πραγματικά τι κάνουμε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να βρίσκεται σε μια πλήρη αντίφαση. Από τη μία πλευρά να θέλει να μειώσει κατά ένα βαθμό Κελσίου τους στόχους της COP21 και από την άλλη να μην δίνει τα χρήματα προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Επομένως, το ποσοστό του 50% θεωρώ ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξο. Είδα ότι υπάρχουν και πολλές σχετικές τροπολογίε και ελπίζω οι συντάκτε των δύο αυτών εκθέσεων να αποδεχθούν και αυτοί αρκετά φιλόδοξοι. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα υποστόχος 20% για την ενεργειακή απόδοση, αν πραγματικά θέλουμε να συνάδουμε κι εμεί με τι απαιτήσει που προβάλλουμε προς τη δική μας την κοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε φορά που προωθούμε τέτοια επενδυτικά σχέδια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να επαναλάβω τα υπευθυμητικά μου σχόλια και την ευγνωμοσύνη μου τους ε, εισηγητές να μιλήσαμε για τους αυτοκινητοδρόμους. Με βάση αυτά που ξέρουμε, σίγουρα έχει εφαρμοστεί το σχέδιο Juncker. Οπότε το ΕΦΣΥ δεν θα πρέπει να αποτελέσει τρόπο για ε, μη εξορθολογισμό των ε, δημοσίων δαπανών και του δημοσίου χρέους. Να, να υπάρξει δηλαδή να έχουμε με αυτόν τον τρόπο ε, σε τόσο ιστορικά χαμηλές ε, τιμές πρόσβαση και να μην χρησιμοποιούνται. Το ΕΦΣΙ λοιπόν ε, σύμφωνα με τόσο λένε οι Δήμοι ας πούμε και οι τοπικές αρχές είναι πράγματα που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να κρίνουμε το FC1 και να μπορέσουμε να ε, οριοθετήσουμε κάπως καλύτερα το FC2. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος τον λόγο, οπότε μπορούμε να δώσουμε τον λόγο στους συνεισηγητές μας. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. Αντίστροφα από ό,τι πριν, ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χρηματοδότηση είπαμε και η Κομισιόν είπε ότι ότι ποτέ ξανά δεν θα παίρναμε χρήματα από τα προγράμματα που είχαμε ήδη πάρει. Πάκτε sunt σερβάντε. Δηλαδή, ούτε από τον ορίζοντα 2020, ούτε από το διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Και αυτό είναι ο λόγος που δεν θέλουμε να πάρουμε τα 500 εκατομμύρια από το Connecting Europe Facility. Τα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε ε, τα παίρνουμε και βάζουμε όλα τα χρήματα στις επιδοτήσεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν η Κομισιόν λοιπόν και τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι αυτά τα 500 εκατομμύρια είναι κάτι φοβέρο για ένα τέτοιο σχέδιο, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Είχαμε αυτά τα 500 εκατομμύρια και τα περιθώρια που ήταν ήδη στην πρόταση της Κομισιόν. Ε, τα 150 εκατομμύρια, συγγνώμη και τα 500 δεν θα τα πάρουμε από προγράμματα που, από, από τα οποία έχουμε πάρει χρήματα. Θα πάρουμε από τα περιθώρια. Νομίζω ότι αυτό είναι λογικό. Δεν πρέπει να αγγίξουμε το Connecting Europe Facility γιατί το έχουμε ήδη αγγίξει. Και αυτό το ποσό δεν είμαι σίγουρος ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο ε, τις επιπτώσεις από την έξοδο της ε, Βρετανίας και για τα περιθώρια. Θα τα χρησιμοποιήσουμε και πρέπει να μιλάμε για δεσμεύσεις και συμβιβασμούς. Πρέπει να τηρούμε το λόγο μας και τις συμφωνίες μας. Είχαμε πει ότι ποτέ ξανά δεν θα πάρουμε χρήματα, επιμένω από το Connecting Europe Facility και από τον ορίζοντα 2020 και ότι πρέπει και πρέπει να σεβαστούμε και τους συμβιβαστισμούς και τις δεσμεύσεις μας. Τώρα για το FC2. Έχει νόημα να μιλάμε γι' αυτό. Είτε το θέλουμε είτε όχι υπάρχει κενό επενδύσεων. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Είτε συμφωνούμε είτε όχι λειτουργεί το ΕΦΣΙ, μπορεί να βελτιωθεί. Αυτός είναι ο στόχος και, μέσα, και στη διάσταση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει σχεδόν ε, εξαντληθεί το κομμάτι των εγγύσεων. Υπάρχει λοιπόν λόγος να συνεχίσει το FC2. Το FC2 πρέπει να πάει μέχρι το 2020, είμαστε στο 2017. Πόσο ε, χρόνο χρειάζονται τα project για να εκτελεστούν. Οι επενδυτές δεν έχουν ανάγκη για προβλεψιμότητα. Υπάρχει λοιπόν νόημα για όσους θέλουν επενδύσεις, απασχόληση και βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχει νόημα και μάλιστα είναι εκτακτή ανάγκη να έχουμε μία πρόταση για να μπορέσουμε να δώσουμε προβλεψιμότητα και για να μπορέσει αυτό το ταμείο να υπάρξει μέχρι το 2020. Γιατί ακούω πολλές φορές σχόλια και παρεμβάσεις που λένε ότι θα πάει μετά το 2020. Όχι, μέχρι τότε είναι η παράταση. Και τις επιπτώσεις θα τις δούμε τώρα. Θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Αν τις περιμένουμε αυτές θα πρέπει να περιμένουμε πάνω από 10-15 χρόνια. Υπάρχουν διάφορες ανησυχίες που συμμερίζομαι από την πλευρά της Κομισιόν. Μιλάω για τη σχέση με τις Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες, NPBs. Ο στόχος δεν είναι να θέσουμε σε κίνδυνο την λογοθεσία, το accountability. Ο στόχος δεν είναι να δημιουργήσουμε γεωγραφική συγκέντρωση και να την προωθήσουμε. Αλήθεια, όντως, αν ενισχύσουμε τους όρους ε, ε, συμμετοχής για αυτές τις ε, τράπεζες, ξέρουμε ποιες θα πάρουν τα χρήματα. Πρέπει όμως να μετριάσουμε αυτή την κατάσταση και να ενθαρρύνουν με τις τράπεζες αυτές ώστε να γίνουν πιο ισχυρές γιατί δεν υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε, να το έχουμε στο μυαλό μας. Επίσης θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε με κάποιον έλεγχο πάντοτε τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες. Πρέπει να τις ευαισθητοποιήσουμε ώστε να επιτύχουν το στόχο να έχουν πλατφόρμες, να μην υπάρχει συγκέντρωση γεωγραφική μέσω αυτών πάντοτε. Και ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε συμβαστική λύση και για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους που έκαναν τις προτάσεις τους και που θέλουν να μπορέσει η Ευρώπη να έχει επενδύσεις σε διαφορετικούς τομείς. Σίγουρα ο στόχος του κλίματος πρέπει να διέπει όλα τα έργα, όλα τα project. Αν έχουμε έναν ενδεικτικό στόχο και μπορέσουμε να τον ξεπεράσουμε ακόμα καλύτερα. Όμως ο στόχος μας και οι πολιτικές μας είναι ξεκάθαρες και είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η ΕΤΕΠ πρέπει να σέβεται και να ερμηνεύει σωστά τον κανονισμό. Θεωρώ ότι η ΕΤΕΠ πρέπει να το κάνει, είναι υποχρεωμένη. Αν ένας αυτοκινητόδρομος γίνει με το ΕΦΣΥ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς αυτό. Αυτό είναι η προσθετικότητα και η σωστή ερμηνεία. Να ενισχύσουμε όμως τα κριτήρια της προσθετικότητας για να είναι πιο ξεκάθαρα. Πρέπει να το προσπαθήσουμε, αλλά ομολόγω και το έχω πει πολλές φορές, δεν ξέρω αν θα είναι τόσο εύκολο να βελτιώσουμε τον ορισμό της προσθετικότητας. Η ερμηνεία πρέπει να είναι σωστή. Κάποιες φορές φοβάμαι ότι όταν προσπαθούμε να βελτιώσουμε νομοθετικά κείμενα, τελικά τα κάνουμε πιο περίπλοκα και συνεχίζουμε να διαονίζουμε το πρόβλημα της ερμηνείας. Και η ερμηνεία της προσθετικότητας, κατά τη γνώμη μου, είναι ξεκάθαρη. Αν μπορούμε να τη βελτιώσουμε, ας το κάνουμε, αλλά και το στόχο του κανονισμού που είναι να βελτιώσουμε ό,τι μπορούμε να βελτιώσουμε για να λειτουργήσει καλύτερα αυτό το ταμείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ούτο Μπούλμαν. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαστε σε μια κατάσταση που θα την συνοψίζαμε ως εξής. Ναι, βλέπουμε ότι δεν έχουμε τόσα σοβαρά προβλήματα στην έκθεση ίδιας πρωτοβουλία και οπωσδήποτε θα μιλήσουν και οι ίδιοι και θα καταλήξουμε νομίζω σε ένα καλό αποτέλεσμα. Στο νομοθετικό τμήμα αναφέρθηκαν ε, τα σημεία τα οποία ανέμενε ο Χωσέ Μανούλ Φερνάντες και η ταπεινότης μου. Ε, Παρ' όλα αυτά, ναι, ξέπληξε το πόσο μεγάλη ήταν η ενότητα στον συνδυασμό αυτών επιτροπών για να προωθήσουμε το ΕΦΣΥ, έχουμε το ίδιο πλαίσιο, τα ίδια σημεία κριτική στις ίδιες ιδέες για το τι θα κάνουμε από εδώ και μπρος μέσω της ε, τράπεζας. Όλες οι ομάδες που μίλησαν οπωσδήποτε δεν θέλουν να υπάρξει κάποια απόθεση ιδιωτικών κονδυλίων μέσω του ΕΦΣΙ, θέλουν την βιωσιμότητα. Ξέρουν ότι το ΕΦΣΙ δεν θα μπορεί να γεμίσει το μεγάλο κενό των επενδύσεων, αλλά θα μπορούσε να κινηθεί με βάση τη λογική της καλύτερης επενδυτικής συμπεριφοράς και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Η ενότητα λοιπόν υπάρχει και η συζήτηση επικεντρώνεται σε τεχνικά ζητήματα. Με ποια μέσα με ποιες βελτιώσεις ε, θα πάμε από το α στο β. Εδώ ήθελα να αναφερθώ στους συναδέλφους ε, που μίλησαν και σε όσους υπέβαλαν γραπτές ε, τροπολογίες και να πω ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να φανεί αυτή η συνένεση και στο κείμενο ή οι συγητές είναι διατεθειμένοι να δεχτούν πολλέ τροπολογίε, να είναι ευέλικτοι για να δώσουν την εντύπωση αυτή και βεβαίως αυτό ισχύει και για τους στόχους του κλίματος που αναφέρθηκαν ρητός, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, κάθε άλλο. Και θα συζητήσουμε οπωσδήποτε ποια είναι η καταλληλότερη μορφή και πού πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Βεβαίως, στον κύριο Σολέ θα ήθελα να πω ναι, καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας δεν υπάρχει κάποια αντίφαση σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπω και στους ε, συναδέλφους. Έχουμε... Ε, δεν θέλουμε εμείς να υπάρχει πουθενά διαφάνεια. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Αν υπάρχει κάποια πρόταση, κάποια λέξη που λείπει, πείτε μας. Ε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς. Κάθε άλλο θέλουμε πλήρη διαφάνεια. Λοιπόν, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, σε επικοδομητικό δρόμο. Ε, επιτρέψατε μου να πω δύο λόγια στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ για τις επικοδομητικές συζητήσεις που είχαμε για την ε, ολοκληρωμένη κριτική των διαφόρων σημείων που αναφέρθηκαν. Ε, οπωσδήποτε θα συνεργαστούμε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κάνω μια παρατήρηση. Την εξή που είναι αν θέλετε και μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Η Κομισιόν λέει ότι θέλει όπως και εμείς ε, περισσότερη διαφάνεια, η φορεία, θέλει να είναι στοχευμένα τα μέτρα και να μην υπάρξει βεβαίως κάποια απόθυση υφιστάμενων επενδύσεων. Όμως η Κομισιόν είναι κατά 50% η αρχή η οποία διευθύνει το ΕΦΣΥ. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει γιατί δεν έχει καταφέρει αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Να το πω δηλαδή αλλιώ. Δεν έχουμε επιτύχει τους στόχους μας για βελτιώσεις και όταν κάνουμε προτάσεις δεν αρκεί τελικά να μας πει η Κομισιόν τι δεν της αρέσει αλλά θα πρέπει να πει σε ποια σημεία θα κάνει κάτι για τις παρατηρήσεις μας και Βεβαίω ε, θα μπορούσε να επιδείξει και κάποια δημιουργική πρωτοβουλία για να λύσει κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε μόνο πως η τιμολόγηση δεν είναι θέμα, η νομική υπηρεσία λέει κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει από την νομική υπηρεσία της Κομισιόν. Στη χρηματοδότηση διαφωνούμε. Junior positions δεν πρέπει να ενισχυθούν. Δηλαδή λέμε παντού όχι. Δεν ξέρω αν ε, η COP21 με την ε, μορφή η οποία προτείνεται είναι τόσο δύσκολη όπως ε, λέτε. Ήδη ένα 35% υπάρχει στο χαρτοφυλάκιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Εντάξει, δεν είναι τεράστιο άλμα προς τα εμπρός. Α, μπορούμε να το ξαναδούμε και εάν δεν θα θέλατε την άμεση διαχείριση των εγγυήσεων από τις Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες, πρέπει να μας εξηγήσετε πώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα έχει ένα πιο ευέλικτο σύστημα. Αλλιώς δεν γίνεται. Και εδώ πέρα υπάρχει μια αντίφαση ε, σε αυτά που λέει η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν μπορεί να λέει ότι πρέπει να εξετάσουμε όλες τις λεπτομέρειες μόνοι μας, αλλιώς δεν υπάρχει δέουσα επιμέλεια και επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν μπορούμε να εγκρίνουμε μικρά και μεσαία έργα. Όχι. Θέλουμε να το λύσουμε αυτό γιατί είναι πρόβλημα ουσίας και αν έχει η Κομισιόν κάποια καλύτερη ιδέα για το πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, καλύτερες ιδέες από τις προτάσεις μας για την τιμολόγηση, καλύτερες ιδέες για τη συμμετοχή περιφερειακών αναπτυξιακών τραπεζών. Ε, να τις καταθέσει αλλά στην νομοθετική αυτή διαδικασία η Κομισιόν δεν μπορεί να περιορίζεται στο να λέει μόνο όχι. Γιατί θέλουμε κάτι καλύτερο και χρειαζόμαστε και τη συνεργασία της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπορούμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε την ε, συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ τους εισηγητές, την ε, Κομισιόν ε, και όσους συμμετείχαν. Η ψηφοφορία στις δύο εκθέσεις θα γίνει την Δευτέρα 24 Απελίου, 3 ώρα τα απόγευμα στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ. Θέλετε τίποτα άλλο? Όχι, λέει τη συνεδρίαση.